μια συνέλευση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ και φτάσαμε στο τέλος της συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι. Η μερίσια διάταξη προβλέπει τώρα τις παρεμβάσεις ενός λεπτού και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζεμπόσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα πως ε, στην περίπτωση που ένας υγιής άνθρωπος θέλει να προχωρήσει σε φανασία θα πρέπει το, να υπάρχουν οι ε, απαραίτητες συνθήκες αλλιώς παραβιάζεται το άρθρο 8. Κατά τα λοιπά το κράτος εγγυάται το δικαίωμα της ζωής σε όλους τους ε, ανθρώπους. Αυτά τα επιβεβαιώνει νομίζω και η κατάσταση ε, ε, που ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όπως και το δικαίωμα στην ε, ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε όλους τους συναδέλφους που αγνοούν ε, το τι είναι μια φυσική οικογένεια. Δηλαδή όταν άνθρωποι που είναι υγιείς ε, θεωρούν πως έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε ευθανασία, μάλλον κάτι επέκαλα. Σας ευχαριστώ κύριε Σπυρίλο. Πρόεδρε, θα ήθελα ενώπιον αυτού του κοινοβουλίου να πω πόσο μου φαίνεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλή τον κύριο Μπαρόζο να υπονομεύσει την υγεία και την ασφάλεια εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά και ταυτόχρονα τους επιβάλλεται λιτότητα. Οι νέοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και να ψάξουν δουλειά αλλού γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Δεν μπορούν ε, οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζονται σε εγκληματίε λόγω των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να σταματήσουν αυτέ οι πολιτικέ ε, τη καταδίκη ε, των πολιτών. Οι πολίτε έχουν στραφεί κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατηγορούν, ενώ το αντίστροφο θα πρέπει να συμβαίνει. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερο κύρο, περισσότερη εξουσία στου Ευρωπαϊκού θεσμού. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε την ασφάλεια, την ανάπτυξη, την υγεία και την ευημερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να του δείξουμε ότι είναι υγιή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματά του. στην ε, μέση της χειρότερης οικονομικής ε, κρίσης που έχει χτυπήσει, τη χειρότερη οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει στην Ιρλανδία, έχουμε δύο ε, ελπίδες στον τομέα των εξαγωγών και της γεωργίας. Η γεωργία όμως πλήττεται λόγω των καιρικών συνθηκών. Ξεκίνησαν αυτές το δεύτερο εξάμεινο του 2012 και συνεχίστηκαν το 2013. Μεγάλα τμήματα της χώρας, ειδικά η περιφέρειά μου, δεν είχαν καθόλου ανάπτυξη των φυτών ε, και πάρα πολλά προβλήματα με τον χώρο. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, χορτάρι για ζωοτροφή και μπορούν τα μπορεί τα προβλήματα να συνεχιστούν και το επόμενο έτος. Υπάρχουν προσπάθειες βοήθειας από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, αλλά τα ζώα ψοφάνε ενώ προσπαθούμε να κάνουμε εισαγωγή ζωοτροφής, ε, αγρότες και ζώα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η κρίση της ζωοτροφής υπολογίζεται πως θα κοστίσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο στους ε, αγρότες μας. Ζητάω λοιπόν από την κυβέρνησή μας να ζητήσει άμεσα βοήθεια από το Ταμείο Λεγγύης για να υπάρξει κάποια ανακούφιση. Ευχαριστώ η κυρία... Η κυρία Νταμαρτίν, ευχαριστώ πρόεδρε ο λιμένας της Γένοβας και το πρόσφατο ατύχημα εκεί όπου έχασαν την, ε, τη ζωή τους 9 άτομα που δούλευαν απλώς στο γραφείο τους είναι κάτι που αποδεικνύει ότι πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή των άλλων. Δεν θα ήταν μοιραίο το ατύχημα αυτό αν είχαν ληφθεί τα απόλυτα κατάλληλα μέτρα. Έπρεπε να έχει αλλάξει σημείο η προσέραξη των μεγάλων καράβιων σε αυτό το λιμάνι εδώ και χρόνια. Δεν έλαβε κανείς μέτρα προστασίας. Δεν έπρεπε να επαγρυπνεί κάποιο να εποπτεύει. Πάντω κανεί δεν το έκανε και κανεί αυτή τη στιγμή δεν είναι ηθικά υπόλογο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο λιμάνι τη Ευρώπη με τεχνικέ προδιαγραφέ που θα έπρεπε να είναι στο ύψο των περιστάσεων. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτική, ε, δεν θα έπρεπε να είναι θέμα μόνο πολιτική επιλογή το ποιο είναι υπεύθυνο σε τέτοιου λιμανιού. Γι' αυτό φέρω το ε, θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αρκεί η έρευνα που θα γίνει σε επίπεδο Ιταλικού κράτου. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμαρτίνη. Τώρα ο κύριο Μπάτ Ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρία της ομάδας που θα γίνει στην Αγγλία. Η τοποθεσία θα είναι το ξενοδοχείο Grove Walkford από τις 6 9 Ιουνίου. Αυτές οι αιτήσιε συναντήσεις είναι σύνοδοι κορυφή των πιο ισχυρών ανθρώπων στον κόσμο της πολιτικής, της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Το μεγάλο μυστήριο περιβάλλει αυτές τις συνεδριάσεις ε, ε, είχαν σαν αποτέλεσμα από το 1994 να μην τις ε, καλύπτουν τα μέσα ενημέρωσης. Το μυστικό όμως έχει πλέον βγει στο φως και όλα τα μέσα ρωτούν, ζητάνε κατά πόσο θα μπορέσουν να καλύψουν αυτή την συνάντηση και αν όχι γιατί καιρό. Ε, θέλουμε και επίση απεύθυνα μία ερώτηση στις αρμόδιες αστυνομικέ αρχές για να μάθω ποιοι θα καλύψουν τα έξοδα για την προστασία εκείνων που θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε κύριος Μάγκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Μιλάμε συχνά για, την, ε, για το σφασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολλοί όμως στην Ισπανία δεν ε, ε, σέβονται τα δικαιώματα αυτά. Μάλιστα υπάρχει απόφαση της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι θεματοφύλακα των συνθηκών και να φροντίζει για το δίκαιο της το εμπράγματο δίκαιο που θα έπρεπε να προστατεύεται και την υλοποίησή του. Στην Ισπανία, στην Ινταλουσία συγκεκριμένα, πέρασε νομοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία όπου πρόσφατα διασφαλίστηκε ότι η δυνατότητα έξωσης δεν θα μπορεί να επιβάλλεται με τις ίδιες ε, προδιαγραφές. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε εάν ήταν δίκαιη η οδηγία για το εμπράγματο δίκαιο του 1993. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπρόνς. οι όροι φιλοευρωπαίος και αντιευρωπαίος ε, χρησιμοποιούνται ε, και για να εννοούμε υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θεωρώ πως ε, ο όρος αντιευρωπαίος για εμάς που είμαστε αντίθετοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσβλητικός. Η Ευρώπη είναι πολύ παλαιότερη και σημαίνει πολύ περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτισμική, μια θρησκευτική οντότητα και μια οντότητα με συγγενικές ε, καταγωγές η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιευρωπαϊκή γιατί οι πολιτικές της τελικά θα καταστρέψουν την ιδιαιτερότητα της Ευρώπης. Αν έρθουν ε, μετανάστες από τον τρίτο κόσμο θα γίνουν Δεν θα γίνουν νέοι Ευρωπαίοι, αναπόφευκτα θα καταστήσουν μέρη της Ευρώπης τρίτο κόσμο. Ο παγκόσμιος καπιταλισμός και οι παρόμοιες ιδεολογίες είναι υπέρ της μετανάστευσης γιατί θεωρούν τα ανθρώπινα όντα μόνο παραγωγικούς συντελεστές. Ο κύριος Νικουλέσκου έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Επιτροπής για αυτή τη δημόσια συζήτηση για τις ε, μεταβολές στην ε, Γενική και Ανατολική Ευρώπη που θα μας δώσει ε, χρήσιμα στοιχεία για να το πώ θα καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Η Ρουμανία, η χώρα που εκπροσωπώ, δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, παρόλο που είναι εκτεθειμένη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. τα, τα, μετρολογικά, τα, μετεωρολογικά φαινόμενα αυξάνονται και τεράστιε εκτάσεις θα απεριμωθούν στη Ρουμανία. Ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμο το αποτέλεσμα αυτής της συζήτηση και θα ωφεληθεί από τα αποτελέσματά της όλη, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια ε, έδειξαν ότι ε, κάποιες διατάξεις του συντάγματος ερμηνεύθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πιο αποτελεσματικό. Η αναθεώρηση του συντάγματος δεν μπορεί να είναι αναθεώρηση που καθοδηγείται από μια πλειοψηφία. Η κυβέρνηση της ε, Ρουμανίας ζήτησε λοιπόν από την Επιτροπή της Βενετίας, όπως συνέβη και με την άλλη αναθεώρηση του 2003, να εξετάσει προσεκτικά το κείμενο που θα θα ετοιμάσει η Συνταγματική Επιτροπή. Διεθνή και κορυφαία ιδρύματα θα εξασφαλίσουν ότι όλα τα στοιχεία, που, όλα τα στοιχεία της αναθεώρησης τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αναθεώρηση του συντάγματος δεν είναι μια ε, εκμετάλλευση της πλειοψηφίας της μειονότητας από την πλειοψηφία. Πρέπει λοιπόν να ετοιμάσουμε ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να ισχύσει για πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον. Ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη. Ο κύριος Πρίξ γεννήθηκε στο Μπάλεν, στην ε, περιφέρειά μου, στην Λονδίνο. Και έχασε το, τη ζωή του όταν το 1982 το Σέφιλντ ε, βυθίστηκε στα νυχτά της Αργεντινής στα Φόκλαντς. Ε, ήταν ε, ένας άνθρωπος ο οποίος έλαβε παράσημο για την ε, τόλμη του και την υπερηφάνειά του προσπαθώντας να σώσει το πλοίο του. Επίσης άλλοι 200 στεκτικοί έχασαν τη ζωή τους και επίσης πολλοί άμαχοι ε, τραυματίστηκαν για να ανακτήσουμε τα Φόκλαντς για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δυστυχώ κρίμα να μην δέχεται το σώμα αυτό, κάτι που και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ορίσει ως υπεράκτια διαμερίσματα. Και είναι κρίμα που τα νήσι Φόκλαντς που ψήφισαν σε δημοψήφισμα υπέρ της παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην μπορούν να επιβάλλουν το δικαίωμά τους αυτό και την άποψή τους. Έτσι λοιπόν για τις 250 οικογένειες που έχασαν ανθρώπους τους πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη ε, ακόμη και, στα μέλη, και στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στους πολίτες των νήσων Φόκλαντ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν είναι βρετανική, ε, βρετανική Φόκλαντ. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Σόζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Την ημέρα που ο κύριος Μπαρόζο δήλωσε ότι η λιτότητα πρέπει να συνεχιστεί στην Πορτογαλία και ότι οι πολιτικές παρόλα αυτά που έχουν επιβληθεί ως τώρα δεν είναι βιώσιμες και δεν είναι αποτελεσματικές, φάνηκε ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική μας πορεία. Βλέπουμε ότι βγουν σε κοινωνική τραγωδία οι πολιτικέ λιτότητα και ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που δημιουργεί ακόμη και περισσότερο ύφεση. Το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Πορτογαλία αποφάσισε πολλά δημοσιονομικά μέτρα ε, και έκρινε πολλά δημοσιονομικά μέτρα τη Τρόικα αντισυνταγματικά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δεσμεύσει του προγράμματο προσαρμογή δεν θα μπορέσουν να τηρηθούν από την Πορτογαλία. Θα πρέπει να μην επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη λιτότητα και την ύφεση. Η άνθρωποι τη Πορτογαλία το κατέλαβαν αυτό και το 82% των πολιτών σε πρόσφατε δημοσιοποιήσει ζητούν την επαναδιαπραγμάτευση ή την υπαναχώρηση τη Τρόικα από τι θέσει τη. Όμω αυτό ακόμη δεν έχει απηχηθεί. Δεν ή θα ήταν μια καλή ιδέα να ακούσουμε επιτέλου αυτό που έχουν να μας πούν οι πολίτες. Ευχαριστούμε κυρία Σόζα. Ο κύριο Μπάνκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το 2013, τον Οκτώβριο του 2013, είναι η τελευταία ημερομηνία της μετάδοσης της οδηγίας για τα δικαιώματα και αυτή η ημερομηνία θα σημάνει την αρχή μιας περίοδου όπου κάθε πολίτης μπορεί να αποφασίσει σε ποια πόλη πρέπει να πάει για να εξασφαλίσει θεραπεία, την απαιτούμενη θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ιαματικά λουτρά πρέπει να αξιολογούνται λοιπόν με το ίδιο σύστημα παντού ε, για να αντιπιστωθεί ότι οι θεραπείες δεν έχουν παρενέργειες και δεν κοστίζουν ε, ε, και κοστίζουν πιο φθηνά από τα σύγχρονα φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να καθιερώσουμε ένα σύστημα βάσει του οποίου η ποιότητα των ιαματικών νερών και οι ιατρικές θεραπείες που παρέχονται εκεί μπορούν να ρυθμίζονται ώστε να αποφασίζουν τι θα κάνουν οι ασθενείς. Ευχαριστούμε κυρία Σαρμπού. Ευχαριστώ. Το 2010 ήμουν συντάκτης και εγώ του ψηφίσματος που απαγορεύει τη χρήση κυανίου στα ορυχεία. Υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επέμεινα και σε άλλες επιστολές και δηλώσεις το ίδιο θέμα και η Κομισιόν είπε πως δεν θέλει να ε, δώσει συνέχεια. Όμως ε, υπάρχει ανησυχία στους Ρουμάνους πολίτες. Αυτή τη στιγμή αναθεωρείται η σχετική νομοθεσία, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιες επικίνδυνες ε, ουσίες. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι όταν μιλάμε για τη χρήση κιανίου στα ορυχεία. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιό να απαγορεύσει αυτές τις ουσίες στην προσοχή μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ. Κύριο Ζαρνέκη, επόμενος ομιλητής. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, już e, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πρόεδρε, ήδη έχουν περάσει τρία χρόνια από την αεροπορική τραγωδία του αεροπλάνου του Προέδρου της Πολωνίας στο Σμόλενσκι και στη Ρώσια. Έχασε τη ζωή του ίδιου και επτά μέλη της ε, πολωνικής πολιτικής ελίτ. Έως σήμερα όμως τα συντρίμια του αεροπλάνου αυτού και το μαύρο κουτί βρίσκονται ακόμη στη ρωσική επικράτεια και δεν έχουν επιστραφεί στην Πολωνία. Η έρευνα για το θέμα αυτό ε, βλέπουμε να διεξάγεται με πάρα πολύ βραδείς ρυθμούς. Υπάρχει λοιπόν η υποψία ότι αυτό γίνεται εκ προθέσεως και μάλιστα λόγω ρωσικών ε, αποφάσεων. Σε διεθνέ λοιπόν επίπεδο πρέπει όλοι να συνεργαστούμε προκειμένου να διαλευκανθεί η Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, στον κύριο Τούσα. Η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της προωθείται με προτεραιότητα την κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση, μαζική ανεργία, φτώχεια για τους εργαζόμενους και ένταση του αυταρχισμού της κρατικής καταστολής και βίας την ποινικοποίηση των εργατικών λαϊκών αγώνων. η αντιλαϊκή πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης τροφοδοτεί τον ρατσισμό και την ξενοφοβία φουσκώνει τα πανιά των φασιστικών ναζιστικών μορφωμάτων. στην ελλάδα η τρικομματική κυβέρνηση νέα δημοκρατία πασόκ δημάρ έχει θέσει υποδιωγμό το δικαίωμα της απεργίας μετά την πολιτική επιστράτευση των αυτεργατών των εργαζομένων στο μετρό στου ο타ε η κυβέρνηση επιστράτευσε τους καθηγητές μέσης εκπαίδευση. το 98 των απεργών κηρύσσονται παράνομε από τα δικαστήρια. την ίδια επίθεση εξαπολύουν οι αστικέ κυβερνήσει σε όλα τα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ισπανία όπου δεκάδε πρωτοπόροι αγωνιστέ μέλη και στελέχη του κομμουνιστικού κόμματο των λαών τη Ισπανία απεργεί στη γαλλία την πορτογαλία και άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωση αντιμετωπίζουν ποινέ φυλάκιση και εξοντωτικά χρηματικά πρόστιμα γιατί συμμετείχαν σε διαδηλώσει και απεργιακέ κινητοποιήσει. στην ελλάδα οι εφοπλιστέ στι 22 μάη σύρουν στα δικαστήρια στελέχη του κομμουνιστικού κόμματο ελλάδα συνδικαλιστέ ναυτεργάτε του παμε ζητώντα του αποζημιώσει εκατομμυρίων ευρώ γιατί υπερασπίστηκαν με απεργιακέ κινητοποιήσει τα δικαιώματα των ναυτεργατών. Ευχαριστούμε κύριε Τούσα. Τώρα κυρία Τούνεν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πρέπει τη Είναι δύσκολο να ε, δούμε ποια είναι η αλήθεια σε ορισμένα ζητήματα. Ο κύριος Σικόρσκι ε, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες ενός συλλόγου, ο οποίος έχει στόχο όχι μόνο να ξεχαρίσει το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην ε, χώρα μας, αλλά και άλλους σκοπούς. Αυτό είναι μόνο ένα σημάδι του ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για την ελευθερία του τύπου και να υποστηρίζουμε πολιτικούς κρατούμενους και πρόσφυγες. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνουμε τον Αγγλή για την οργάνωση αυτή για να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Πρόκειται για μια ένωση που αξίζει πραγματικά να υποστηριχθεί γιατί μας δείχνει πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν. Λάσεντερ. Πρόεδρε, μόλις θέλω να καταγγείλω πώς το Λαϊκό Κόμμα επιτίθεται κατά της υγείας, της απασχόλησης και του πολιτισμού ένα θέμα που προβληματίζει, μας προβληματίζει και μας απασχολεί γιατί μιλάμε για ε, επίθεση ε, ε, εκείνων που μιλάνε καταναλυνικά, μια γλώσσα που είναι πλέον διεθνώς αποδεκτή. Η υιοθέτηση νέων κανόνων οδήγησε στη χρήση δύο επιπλέον γραμμάτων. Γι' αυτό θα, ήθελα να καταδικάσετε και πάλι όπως το κάναμε ήδη ως μέλη της ομάδας των μειονοτικών γλωσσών. Μιλάμε για ένα θεμελιώδες σφάλμα και θα έπρεπε στην Αραγωνία να μπορεί, να μπορεί κανείς να μιλάει τη γλώσσα της χώρας. Ο κύριος Αγκουράκης. Τη στιγμή που σημειώνεται τεράστια συσσόρευση πλούτου και ανάγκες των εργαζομένων συνεχώς αυξάνουν, τα μονοπόλια Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις εντείνουν σε απίστευτο βαθμό την εκμετάλλευσή τους. Σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν την κατάργηση των εθνικών γενικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη λευκή βίβλο του 2012 της Επιτροπής για τις συντάξεις που προβλέπει αύξηση των ορίων ηλικιακής συνταξιοδότησης χτύπημα του δημοσίου χαρακτήρα των συστημάτων ασφάλισης μετατροπή των συντάξεων σε επιδόματα πρόνοιας μετατόπιση των ασφαλιστικών βαρών κράτους και μονοπωλιακών ομίλων στις πλάτες των ασφαλισμένων αξιοποίηση της ασφάλισης ως νέο χρυσοφόρο πεδίο κερδοφορίας. Στην Ελλάδα από την 1η Γενάρη 2015 καθιερώνεται η βασική σύνταξη των 360 ευρώ που δεν αντιστοιχεί ούτε σε επίδομα φτωχοκομείου και αυτό ακόμα το εξευτελιστικό βοήθημα η κυβέρνηση μπορεί να το μειώσει για τη διάσωση τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση απαιτείται η συμπόρευση τη εργατική τάξη και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων με το κομμουνιστικό κόμμα και το εργατικό λαϊκό κίνημα ενάντια στην ευρωπαϊκή ένωση και στο καπιταλιστικό σύστημα για υποχρεωτική καθολική κοινωνική ασφάλιση με εισφορέ που θα βαρύνουν το κράτο και του καπιταλιστέ αξιοπρεπεί συντάξει δωρεάν υψηλή ποιότητα παροχέ υγεία περίθαλψη και πρόνοια. Merci Νίμπλερ, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πολυγλωσία είναι ένας ε, μεγάλος ε, θησαυρό ε, στην Ένωση, αντικατοπτρίζει πραγματικά την πολιτισμική και γλωσσική ε, ποικιλία που υπάρχει στην Ένωση. Πρέπει πραγματικά να κάνουμε περικοπές, ε, το αναγνωρίζω, αλλά πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι στο Κοινοβούλιο. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να καταργήσουν κάποιες συγκεκριμένες γλώσσες. Και τώρα στην Επιτροπή των ε, Περιφερειών λένε πως θα πρέπει να καταργηθούν κάποιες γλώσσες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27 ε, προς 28 κράτη-μέλη και 23 επίσημες γλώσσες. Καμία γλώσσα δεν πρέπει να θεωρείται ανώτερη από άλλες. Ε, συμφωνώ με το ότι πρέπει να γίνουν οικονομίες, αλλά χωρίς να τίθεσε σε κίνδυνο η δημοκρατία και η ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Μίτση, που λαμβάνει για πρώτη φορά τον λόγο. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι και τιμή που είμαι η πρώτη γυναίκα από τη Μάλτα που εξελέγει ως μέλος αυτού του σημαντικού θεσμικού οργάνου είναι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη το Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε στο πλευρό τους και ότι το Κοινοβούλιο θα εξασφαλίσει ότι ε, θα περάσει το ταχύτερο δυνατό αυτή η δύσκολο περίοδο. Δουλεύω στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να συνέλθει από την κρίση η Ευρώπη το ταχύτερο δυνατό. Για να το επιτευχθεί αυτό πρέπει να φροντίσουμε να μην καταστρέψουμε τις οικονομίες μας με υπερβολικά μέτρα λιτότητας και να εστιαστούμε σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι προνόμιο για μένα που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να υπηρετήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους πολίτες της Μάλτας. Υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξω τα συμφέροντα των Μαλτέζων αλλά και των υπολείπων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με όλο το σεβασμό που οφείλω σε αυτό το Ίδρυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μίτση. Πρώτη φορά που λάβατε το λόγο στο σώμα. Η κυρία Νίμπλερ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της απαγόρευσης ε, του ελαιολάδου σε ανοιχτά δοχεία στα εστιατόρια. Εμφανίστηκε στο γερμανικό τύπο ότι δεν θα επιτρέπεται στο μέλλον κάτι τέτοιο. Και απο πρώτης Πρώτου, λέει, 2014 θα ισχύσει αυτή η απαγόρευση σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ανοιχτά ε, ελαιοδοχεία θα απαγορεύονται το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι συνεχώς ε, σε σφραγισμένες συσκευασίες που δεν θα μπορούν να ξαναγεμίσουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο ερώτημα το εάν θα ακολουθήσει και κάτι για το ξύδι και το αλατοπίπερο απάντησε ο εκπρόσωπος Κομισιόν πως ε, πιθανόν να γίνει και κάτι τέτοιο. Ε, ειλικρινά θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν τι άλλο θα α, τους απασχολήσει αντί να ασχολούνται με τα σοβαρά προβλήματα των ανθρώπων να ασχολούνται με το πώς έρχεται το ελαιόλαδο στο τραπέζι. Ε, ζήτω η γραφειοκρατία δηλαδή. Πείτε τα εκεί που θα πάτε στην Κομισιόν κυρία Επίτροπε. Ευχαριστούμε κυρία Νίμπλερ. Και τώρα... Χάθηκα. Απόν, απούσα, απόν. Η κυρία Σμάλκοβα. poslanci, ktorí sa rozhodnú opäť kandidovať. ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, βουλευτές οι οποίοι θέλουν να κατέβουν υποψήφοι θα έχουν να απαντήσουν δύσκολες ερωτήσεις. Στην δε ημέρα της Ευρώπης ε, συναντήσαμε ανθρώπους στους δρόμους οι οποίοι έχουν την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο μία ένωση ε, όταν τα πράγματα πάνε καλά, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν ε, δεν μπορεί να βοηθήσει τους νέους να βρουν δουλειά. Αυτό πρέπει να λάβουμε γρήγορα και όταν ορίζουμε προπολογισμό για τα επόμενα έτη δεν πρέπει να ξεχνάμε τους νέους προγράμματα όπως το Εράσμος και το Γαλιλαίο κτλ. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Κλέβα. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Κλέβα και ακούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο όταν ε, συζητούσαμε το Sixpack δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράσινο φως και της αναθέσαμε το καθήκον να υλοποιήσει τα μακροοικονομικά μέτρα και τους σχετικούς δείκτες. Ε, μέτρα και δείκτες που θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σχετικές συστάσεις προς τα κατημέρια. Υπό το φως της κατάστασης στην χώρα μου και όσων είχε αποφασίσει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θυμίσω ότι οι μακροοικονομικέ ανισορροπίε στην Ευρώπη και η ανάλυση του θα πρέπει να συνάδει με τον κατάλογο των μακροοικονομικών δικτών. Υπάρχει ακόμα μεγάλη κερδοσκοπία από πολλά κερδοσκοπικά funds. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιωθεί ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες ισχύουν. Ευχαριστούμε. Κύριε Γκουτιέρες έχει το λόγο δεν είναι εδώ. Ο κύριος Ταμπάσντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο, οι εκπρόσωποι της οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικό ε, ποσοστό ΦΠΑ για βασικά προϊόντα. Ενώ στην Ουγγαρία το ΦΠΑ είναι 27%. Το υψηλότερο ποσοστό στην ε, Ευρώπη, ενώ στην Αυστρία και στην Πολωνία το ΦΠΑ είναι πολύ χαμηλότερος. Με βάση το, το, το παράδειγμα της Πολωνίας θα αποφασίσαμε να μειώσουμε στο 5% το ΦΠΑ για τα είδη διατροφής, διότι ένα υψηλό ποσοστό ΦΠΑ θα οδηγήσει σε μαύρη αγορά και δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη της ε, γεωργίας ε, στη χώρα. Πρέπει επίσης να μειωθεί, να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των κατοίκων, οι οποίοι χρειάζονται σαφώς σημαντική Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye ή των παρεμβάσεων ενός λεπτού. Θα πρέπει να διακόψω τη συνεδρίαση έως... Η των παρεμβασεων ενό λεπτου θα πρεπει Κορνέλη, η κυρία Κορνέλη όμως ηρθε οπότε... Θα δούμε τι γίνεται με τη δική της έκθεση, παρουσίαση του δικαιωμάτων των γενικών σε 56 Παρακαλώ, καθίστε και έχετε το λόγο. Κυρία Κονέλη, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Και μόλις ε, έρχομαι από ψηφοφορία και με συγχωρείτε για την